Dear colleagues. Señoras y señores. Κυρίες και κύριοι. Please be seated. Be seated and try to... Καθίστε, καθίστε σας παρακαλώ και να προσπαθήσετε να είστε σιωπηλοί. Λοιπόν, όπως είπα, έχουμε τρία έκθεσεις. Για ψηφοφορία πολύ πολύ πλοκά. που θα καταναλώσουν πολύ χρόνο. Καταρχήν, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να συνεργαστείτε για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες με αυτό το τόσο πολύπλοκο θέμα και να μας βοηθήσετε να προχωρήσουμε και να μην υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την ε, απογραφή όταν υπάρχουν δηλαδή κάποιες τροπολογίες που έπρεπε να καταπέσουν γιατί έχουν συμβηθεί κάποιο συμβασμό κλπ. Σας παρακαλώ να συνεργαστείτε μαζί μας εδώ στο Προεδρείο, γιατί είναι δύσκολη η διαδικασία ψηφοφορία. Ίσως η χειρότερη ποτέ που έχουμε ζήσει. Πρωτού την ψηφοφορία μας θα ήθελα να συγχαρώ τους Ιταλούς συναδέλφους που γιορτάζουν η εκατοστή πεντηκοστή επέτειο της του Ιταλικού κράτους. Σας συγχαίρω λοιπόν για την επέτειο αυτή. Σα ε, σας υπενθυμίζω ότι έχετε όλοι τις κάρτες ψηφοφορίας. Ξέρετε ότι κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πρέπει να φροντίσετε λοιπόν να είναι σωστά τοποθετημένη η κάρτα σας. Αρχίζουμε λοιπόν. Παρακαλώ η κυρία Ενφέλ. Μάλιστα σας ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν θέλω να το ζητήσω ενώπιον της Επιτρόπου, αλλά μπορείτε να έχουμε μία γραπτή δήλωση από εσά για το τι σημαίνει ε, συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών. Ναι, ναι, ναι, ναι. Πρέπει να το συζητήσουμε γιατί εμείς ακολουθούσαμε μια συνήθη διαδικασία για τη συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών. Ορισμένε άλλε επιτροπέ αποφάσισαν να συμμετέχουν και οι βοηθοί, δεν ξέρω. Όχι, πρόεδρε, λέει η κυρία Εντφέλη, εγώ δεν αφαιρόμουν στους βοηθού αλλά σε άτομα που δεν έχουν καμία σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει η συνεδρία σε αυτή να γίνει και κλεισμένα των θυρών, αλλά την επόμενη φορά να ξέρω ποιο μπορεί να είναι παρόν και ποιο όχι. Τώρα άντρο. Ναι, ναι, θα φροντίσουμε. Αλλά δεν νομίζω ότι οσδήποτε είναι παρόν εδώ δεν έχει καμία σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά εντάξει, θα δούμε, θα το εξετάσουμε. Άμα έχουμε συνέδρια και κλεισμένων των θερών, θα πρέπει να είναι και κλεισμένων των θερών. δεν έχει κανένα νόημα. Ωραία. Πρώτη ψηφοφορία. Πρόταση δικαιώματο ενημέρωση στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. Η συγγήτρια είναι η κυρία Μπίργκιτ Σίπελ. Αρχίζουμε την ψηφοφορία. Συμβαστική τροπολογία υπερθμών 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Υπέρ. Κυρία Φλότρο. Η δεύτερη παράγραφος ε, της τροπολογίας 139 δεν καλύπτεται από τον συμβιβασμό, άρα πρέπει να ψηφιστεί. Μιλάτε για την δεύτερη συμβιβαστική τροπολογία. Τα criminal proceedings. Α, α, σφάλατε, δεν ήταν για την έκθεση Ζήπερ. Συνεχίζουμε λοιπόν. Συμβαστική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Έχουμε κατά τμήματα ψηφοφορίες. Πρώτη. Η πρόσβαση στα αποδεκτικά στοιχεία κλπ. Το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Εποχές. Για να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. I think it was rejected, but let... Απερίθη, μάλλον, για να είμαστε σίγουροι. The vote is open. Excuse me, split vote. Split vote, compromise amendment. Πρώτα τμήμα της ε, τροπολογίας 3 έχει έξι τμήματα η συμβαστική τροπολογία αυτή. Τρία. Η κυρία Ζήπελ. Να είναι σαφές για όλους τι ψηφίζουμε. Αν ψηφίσουμε κατά τμήματα, αν υπερψηφίσουμε, σημαίνει ότι διατηρείται το τμήμα αυτό. Αν πούμε όχι, απορρίπτεται. Εντάξει, για να είναι σαφές. Now let's proceed. Split first. Λοιπόν, πρώτο τμήμα της συμβαστικής, ηλεκτρονικός έλεγχος για το πρώτο τμήμα. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορία. 28. κατά απερίφθη λοιπόν. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Με την ίδια πλειοψηφία. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται νομίζω. Τρίτο. Τέταρτο, συγγνώμη, υπέρ. Κατά. Αποχές. Το ίδιο, απορρίπτεται. Πέμπτο, με προφορική τροπολογία. Τη άλτε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία Άλμπρεχτ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και γενική ψηφοφορία για την ε, Συμβασική τροπολογία 3. Ηλεκτρονικά. Θέλετε να ελέγξετε την ε, προφορική τροπολογία Albrecht, Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Λοιπόν, προφορική τροπολογία Albrecht, Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. closed. 31 against 19 is Λοιπόν, 31 υπέρ 19 κατά εγκρίνεται λοιπόν πράγματι. Τώρα το σύνολο της τροπολογίας 3. Όπως τροποποιήθηκε. Συμβαστική τροπολογία 3 όπως τροποποιήθηκε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Λοιπόν. Περνάμε τώρα την τροπολογία 55 Λάτφορντ. Όταν εφαρμόζονται αυτά τα δικαιώματα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται νομίζω. Όχι. Να ελέγξουμε. 55 Λάτφορντ το πρώτο τμήμα. Πέρασε. Ναι, είναι κρίθη. Μικρή διαφορά, είναι κρίθη, 25 προς 23. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 61. Ξεχωριστή ψηφοφορία όσο εφαρμόζεται ο εθνικός νόμος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Αυτό απερίφθη. Για να δούμε τώρα. Τροπολογία 75. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πολλές καταπέφτουν και περνάμε συμβαστική 4. Έχει ζητηθεί κατά τμήματα ψηφοφορία από τον κύριο Λέρφορντ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και το σύνολο της συμβαστικής 4, όπως τροποποιήθηκε, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 78. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε. 78. Ελέγχουμε την 78. Η 76 κατέπεσε. Α, δεν χρειάζεται έλεγχος. Ωραία. 79. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στην συμβαστική τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5, ε, 5, συγγνώμη, 5, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6. Με ξεχωριστή ψηφοφορία για το 6-3β. Αυτό ψηφίζουμε ξεχωριστά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το σύνολο συμβαστική 6, όπως τροποποιήθηκε, υπέρ. κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και περνάμε. Συμβαστική τροπολογία 7. Έχουμε μια προφορική Τροπολογία Λάντφερτ. Θα ψηφίσουμε πρώτα αυτή η τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Την συμβαστική τροπολογία 7 ως τροποποιήθηκε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται επίσης έτσι νομίζω όχι να ελέγξουμε 104 104. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 104. Now, the vote is closed. Πέρασε φορές. Ναι, απερίφθη. 38 κατά 12 υπέρ. Περνάμε τώρα στην 108. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 112 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 114. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι δεν ρίχθη. Τροπολογία 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 115 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 116 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβεστική 10 κατά τμήματα ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα της κυρίας Λάτφορντ. It stands. It stands. We're voting on the split vote. Ναι, κατά τμήματα ψηφοφορία. Παρέμβαση εκτός μικροφόνου, Σηκώς υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Λυπούμε, λέει Λάτφορντ. Συμβαστική τροπολογία 10 τροποποιήθηκε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε τώρα that leads us to amendment 125. Τροπολογία 125 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 11. Κατά τμήματα ψηφοφορία συζητήσει λέει δηλαδή υπέρ του τμήματο. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται νομίζω. Τροποποιημένη συμβαστική τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τουρκολογία 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Όχι. Να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε. Την 36. άκρη ψηφοφορία. Board is Πέρασε ψηφοφορίες. Ναι, ναι, είναι κρίθη. 28 προς 23. 137. 137. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στις παραθέσεις και τις γλυκές σκέψεις. Τροπολογία 26. Υπέρ. Κατά. Απαχές. Απορρίπτεται. 28. Υπέρ. Κατά. Απαχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 12. Πάλι με ξεχωριστή ψηφοφορία έχει στήσει η κυρία Λάτφορντ. Πρώτα αυτή, υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απερίπτεται, Συγγνώμη, συγγνώμη. Α, όχι, εγκρίνεται. Η ίδια η κυρία Λάτφορντ καταψήφισε. Αυτό θέλω να πω. Γενικά η ψηφοφορία ήταν θετική. Η κυρία Λέτφορ καταψήφισε. Τώρα έχουμε το σύνολό της συμβαστικής τροπολογίας 12 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 30. Υπέρ. Υπέρ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρέπτεται. Συμβαστική τροπολογία 15. Πάλι με ξεχωριστή ψηφοφορία από τη Lady Λάτφορτ. του υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Λυπούμε κύριε Λάτφορτ. Το σύνολο της τροποποιημένης 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 37 σε δύο τμήματα. 37 όσο έχει υποβληθεί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίφθη. Να. Να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε. Όχι, όχι, απερίφθη. Ναι, παρακαλώ μπορείτε να ελέγξετε και να μας εξηγήσετε γιατί ψηφίσαμε πρώτα το όσο έχει υποβληθεί και μετά κατά τμήματα ψηφοφορία. Αντί αντίθετα, όπως λέει ο δικός μου κατάλογος της ψηφοφορίας. Ε, ο δικός μου λέει άλλα όμως. Συμβαίνει. Συμβαίνει. Ναι. πρώτο stable και μετά όσοι έχει υποβληθεί δηλαδή και μετά το άλλο. Λοιπόν, καταρχήν ψηφίζουμε την τροπολογία 37 χωρίς όσο είναι δυνατόν. Χωρίς τη διατύπωση όσο είναι δυνατόν. Διαφωνεί κανένας. Μα νομίζω ότι θα ήταν ξεκάθαρο να ψηφίσουμε μόνο αυτή τη διατύπωση. Ωραία. Μόνο αυτή τη διατύπωση και μετά το υπόλοιπο. Α, ναι, ωραία. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε μόνο σε αυτή την διατύπωση. Πρώτα θα ψηφίσουμε την τροπολογία χωρίς αυτές τις λέξεις. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα θα ψηφίσουμε ως έχει υποβληθεί, δηλαδή με αυτή τη διατύπωση. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να αλλάξουμε. Να αλλάξουμε. 37. Now the vote is closed. Πέρασε η φορέα. Ναι, εγκρίθηκε λοιπόν. Εγκρίθηκε. Περνάμε τώρα στη 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 44 υπέρ κατά αποχές δεν είδα δεν τα ξεκάθαρα για να ελέγξουμε 44 για να ελέγξουμε Άρχιψη ψηφορία 44 Πέρασε. Εγκρίνεται. Δεν είχα σηκώσει τα χέρια μου στη σοσιαλιστική ομάδα, γι' αυτό δεν σας είδα ξεκάθαρα. Λοιπόν, 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ. The vote is open. The vote is closed. Άρχισε η ψηφοφορία. Πέρας τώρα, ναι. Εγκρίνει ναι, υπέρ και τρεις κατά. Συγχαρητήρια κύριε Ζήπερ. Moving on to the second voting list which is a not less important dossier. We're having an orientation vote. Λοιπόν, ε, έχουμε τώρα την επόμενη έκθεση του κυρίου Σιμών Μπουσουτήλ για την Frontex. Ας ξεκινήσουμε. This is going to be a little complicated, so I, I, I ask for indulgence beforehand. <laughs> Let's go ahead. Λοιπόν, επειδή θα είναι πολύ περίπλοκη οι ψηφορία, παρακαλώ να συγκεντρωθείτε. Συμβαστική 1. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και 1-3-1 ε, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 209. Υπέρ. κατά αποχές νομίζω απορρίφθηκε Πάμε τώρα στη συμβαστική 4 ε, σε τμήματα. Θα ψηφίσουμε σε πέντε τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρίτο, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τέταρτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και πέμπτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα λοιπόν πάμε στη συμβαστική παριθμών 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2-1-2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 7 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 1.03 σε τρία τμήματα ψηφί. Πρώτο τμήμα υπέρ νομίζω απορρίφθηκε δεύτερο τμήμα δεύτερο τμήμα του 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και δεύτερο τμήμα του 103 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 1.05 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Τροπολογία 4 προφορική παρακαλώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 1.07 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Να κάνουμε όμως καλύτερα ηλεκτρονικό έλεγχο. Ελέγχουμε την 107. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 107 και άρχεται η ψηφορία. Ψηφίζουμε. Έκλεισε. Εγκρίθηκε. Μπορεί να, θα πρέπει ίσως να σηκώνετε ψηλά τα χέρια για να βλέπω. Πάμε στην 109. Υπέρ. κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε. Στην 7, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 8, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 9, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται η 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 9 υπέρ αφέτενε κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 112. Μισό λεπτό να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 111. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 111. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφορία. Η 112 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 13, 113 υπέρ κατά απορρίπτεται. Η 114 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Ε, η τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές νομίζω εγκρίθηκε να ελέγξουμε λιγάκι το 10 τη 10 την τροπολογία ε, παρακαλώ ελέγχουμε την τροπολογία υπαρθμών 10 ε, ψηφίζουμε έκλεισε ψηφοφορία εγκρίθηκε Πάμε τώρα στην 115. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πάμε στην 116. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 117. Αποσύρθηκε. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Μισό λεπτό εγκρίθηκε λέει ο πρόεδρος. 119. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Νομίζω εγκρίθηκε, αλλά αν θέλετε να ελέγξουμε, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ελέγχουμε την 119. Ε, ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφορία. Εγκρίθηκε. Προχωράμε. 120. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 121. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 125. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία. 14 και 16. Ε, ψηφίζουμε και για τους υποκοινού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Παράγραφος 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Γκρίνεται. 128. Ε, ε, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ε, αφέτ 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15 παράγραφος 2 ε, υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υποπαράγραφος 2α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 129 μισό λεπτό. Υπάρχει μία υποπαράγραφος 3, ε, τροπολογία 15 υποπαράγραφος 3 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 129 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 130 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 131 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 133 υπέρ κατά αποχές Withdrawn true. Then moving to AFET 12. Favor? 12. Πάμε στο 12, στο άφετ 12, υπέρ κατά αποχές, απορρίπτεται 15, παράγραφος 5, υποπαράγραφος 5, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 135, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, εγκρίθηκε. 137. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 138. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 9 υπέρ. Κατά. απόχέ, εγκρίνεται. Μερικέ έχουν καταπέσει. 145 υπέρ. Κατά. απόχέ. εγκρίνεται. 19 έχει καταπέσει. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άφετ 14 υπέρ Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές, θα ελέγξουμε. 14 ελέγχουμε. 14 αρχίζει, άφετ 14, πέρας ψηφοφορίας. 26 υπέρ, 23 κατά, εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 146 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 147 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 148 υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται. Άφετ 15 έχει καταπέσει διότι εγκρίθηκε η προηγούμενη τροπολογία. Πάμε στην 23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 150 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Άφετ 16 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 149 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 151, 152 έχει καταπέσει, υπέρ της 151, κατά αποχές απορρίπτεται. 153, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 154 με την προφορική τροπολογία του κυρίου Ραμπρινίδη. Υπέρ της 154 κατά αποχές εγκρίνεται. 120 άφετ έχει καταπέσει. Άφετ 17. Άφετ 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 156 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 158 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 159 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 <coughs> υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 160 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται προφορική τροπολογία των πρασίνων γιατί είναι 160 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 162 Α, να ελέγξουμε την προφορική τροπολογία. Ωραία. Ελέγχουμε την προηγούμενη προφορική τροπολογία των πρασίνων και αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 162. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 161 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 163 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 166 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 165 υπέρ Α, έχει καταπέσει, έχει καταπέσει. Ωραία. 32 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 167 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 168 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 169 υπέρ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 Για την 173 λοιπόν αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 29-23 το σκορ εγκρίνεται. 172 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 174 χωριστή ψηφοφορία το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 43 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε εγκρίνεται, εγκρίνεται διορθώνει το πρόεδρος 175 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 176 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται άφετ 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 177 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 178 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 180 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 181 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 183 υπέρ κατά τα αποχές απορρίπτεται 185 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 185 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 186 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι πέρασε. Να το ελέγξουμε. Είχαμε πολλές αποχές, αλλά νομίζω ότι πέρασε. Η 186 λοιπόν, ηλεκτρονικά. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Συνεχίζουμε. 187 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρι... Απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ 48 φωνάζουν όλοι στον πρόεδρο. Συγγνώμη 48. Δίκιο έχετε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 188 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 189 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 50, έχει πέσει 50, κατά πέσει 50, 191 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αν δεν έχει καταπέσει 190, μάλιστα, μάλιστα, 190 λοιπόν, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 195 κυρία Σίπελ έχει καταπέσει. Α, έχει καταπέσει 195, ωραία. Παραμένει έχει καταπέσει. Όχι. Okay, okay. Then we move into 197. 197. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 196 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 198 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 199 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίφθηκε άφετ 26 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 201 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Άφετη 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Είδα ότι μόνο το ΕΛ καταψήφισε. Δεν κάνω λάθος, ε. Να το ελέγξουμε, άντε να το ελέγξουμε. Για την άφετη 27. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Ναι, πέρασε. Εγκρίνεται. 200. Έχουμε, σε, την ψηφίζουμε σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 55, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 202 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 203 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 204 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 205 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 206 υπέρ 206 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 207 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 208 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε απορρίφθηκε είδαμε τι ψήφισε το ΕΛΚΑ ας το ελέγξουμε τέλος πάντων είδα το ΕΛΚ να καταψηφίζει αλλά ας το ελέγξουμε 58 58 Αρχίζει η ψηφοφορία. 58 πέρα της ψηφοφορία. Ε, πέρασε, εγκρίθηκε. Κατά αποχές απορρίπτεται. 230. Συγγνώμη, 213 υπέρ κατά αποχές. 216 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 216. Μα μόλις την ψηφίσαμε τη 216. Α, 215, ναι. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 214 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εξήντα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. εξήντα ένα υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε Εξήντα ένα εγκρίθηκε Άφετη 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 219 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 218 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 218. Λοιπόν, το πρωτότυπο, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 226 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 227 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 31 της άφετ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 228 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 231 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται άφε 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 232 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 233 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 234 με την προφορική τροπολογία αλλά έχει καταπέσει 235 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 236 υπέρ κατά κατά αποχές εγκρίνεται. 37, 237 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 34 της άφετ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 238 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 239 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 241 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται λοιπόν έχει καταπέσει α 63 δεν έχει καταπέσει 63 λοιπόν υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 244 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 245 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 246 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 247 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 248 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 250 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 251 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 68 υπέρ κατά αποχές Εγκρίν. 252 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 254 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Άφετ 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 253 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται λοιπόν ψηφίζουμε τώρα τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 και 74 είναι ίδιες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άφετ 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται λόγω των αποχών φαντάζομαι. Κάνω λάθος αλήθεια. Πολλές φορές δεν βλέπω καθόλου χέρια. Και προσπαθώ να μετρήσω μέσω των συντονιστών αν σήκωσαν το χέρι τους ή όχι. Λοιπόν, άφετ 1. Ελέγχουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άφετ 2 υπέρ. Κατά. Άφετ 2 υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται. Απορρίφθηκε Να το ελέγξουμε. Άφετ 2. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άθε 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να το ελέγξουμε. Μου φάνηκε να κατάλαβα ότι οι φιλελεύθεροι ψήψαν, αλλά ας το ελέγξουμε. Άφετ 3 λοιπόν. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. απορρίπτεται με μία ψήφο. Τέλος πάντων κάναμε ένα λάθος. 80 υπέρ. Τροπολογία 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άφε 4 Α, να ελέγξουμε, να ελέγξουμε την 80. Ωραία, θα ελέγξουμε την 80. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Άφε 4. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2 υπέρ κατά εγκρίνεται. 86 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Προφορική τροπολογία των πρασίνων. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. Άφετ 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 95. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 94. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 97. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 96. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 98. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άφετε 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 99. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τώρα ψηφίζουμε το, το νομοθετικό ψήφισμα και ψηφίζουμε μερικές παραγράφους Τροπολογία 69. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 70 έχει καταπέσει. 71. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το κείμενο τροποποιήθηκε, Υπέρ. Κατά. Δίκιο έχετε, δίκιο έχετε. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία γιατί είναι η τελική ψηφοφορία. Λοιπόν, πέρας ψηφοφορία. Σαραντατρεις, ε, σαραντατέσσερις, σαραντατρεις υπέρ. Ε, κύριε Μπουζουτήλ. Ε, θα ήθελα να μου δώσετε το λόγο για να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω και τους δύο συγκεκριτές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε, να ευχαριστήσω κυρίως ε, τους συμβούλους, ε, τους βοηθούς μου και κυρίως την κυρία που κάθε δίπλα σας, η οποία πραγματικά κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Ευχαριστούμε λοιπόν τις υπηρεσίες γιατί και τους συμβούλους πραγματικά δεν ήταν εύκολη η δουλειά. Πάντως δεν τελειώσαμε ακόμα. Δεν τελειώσαμε. Ε, έχουμε και την τρίτη ψηφοφορία. Τρίτη ψηφοφορία παρακαλώ. Και αυτή είναι αρκετά δύσκολη, φορτωμένη. Σας παρακαλώ λοιπόν ε, να επιδείξετε και πάλι πνεύμα συνεργασίας. Δεν ε, τελειώσαμε. Βλέπω η κυρία Χολμάιερ θέλει να το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα ευθύς εξ αρχής ε, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τους ε, συνεισηγητές μου για το ότι πράγματι σε πολύ δύσκολα θέματα, ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες, παραμείναμε ενωμένοι. Όσον αφορά λοιπόν αυτό το θέμα, το θέμα της μετανάστευσης, αυτό που θεωρώ πολύ σημαντικό είναι ε, να επιτύχουμε όσο δυνατόν μεγαλύτερη συμφωνία και πλειοψηφία. Δυστυχώς δεν έφτασε ο χρόνος έτσι ώστε σε ορισμένα δύσκολα θέματα να βρούμε κοινό παρανομοστή. Θα λοιπόν από πλευράς του ΕΛΚ να πω ότι ανεξάρτητα με το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα ε, θα το έβρισκα πολύ σημαντικό σε αυτά τα δύο-τρία θέματα να επιτύχουμε μεγάλη πλειοψηφία. Γιατί όσο μεγαλύτερη η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο θέμα αυτό τόσο καλύτερη θα είναι και η παρουσία μας απέναντι στο Συμβούλιο και τόσο καλύτερα θα θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και το θέμα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας πω ότι το ΕΛΚ είναι πρόθυμο να διαπραγματευτεί περαιτέρω για ορισμένα θέματα επί των οποίων διαφωνήσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ε, παρατηρήσεις ε, κυρία Χολμάια. Και όπως ε, σας είπα, προχωράμε τώρα στην τρίτη αυτή ψηφοφορία που είναι αρκετά σκληρή και δύσκολη και έχω να κάνω και κάποιες ε, ε, παρατηρήσεις ε, πριν προχωρήσουμε και θα ήθελα και άλλοι να με καταλάβετε γιατί και εγώ κουράστηκα και να σκέφτομαι και να μιλάω. Έχουμε λοιπόν κάποιες παρατηρήσεις. Καταρχήν, να σας πω το εξή Υπήρξαν κάποιες αλλαγές της τελευταίας στιγμής, μα πραγματικά πολύ της τελευταίας στιγμής, λίγες ώρες πριν από την ψηφοφορία. Και θα ήθελα να γνωρίζετε ότι η εισηγήτρια είναι υπέρ της τροπολογίας 109. Δεύτερον, η τροπολογία υπαριθμών 43 καταπίπτει εάν οι 251 και οι 252 εγκριθούν. Τρίτον, οι ακόλουθες ε, τροπολογίες αποσύρθηκαν. Οι 85, 256, 238, 280 και 272. Η κυρία Χίρς ε, κατέθεσε προφορική τροπολογία για τον συμβασμό 10 άρθρο υπαριθμών 38. Θέλετε να λάβετε το λόγο, παρακαλώ. Ε, σύντομα και διαδικαστικό. Όταν ε, θα φτάνουμε ε, στην κάθε φορά στην τροπολογία για την οποία μιλάτε, γιατί δεν το λέτε τότε, γιατί τώρα δεν μπορούμε να τα σημειώσουμε, καλύτερα να τα πείτε όταν θα φτάνουμε στην εκάστοτε τροπολογία, να μας ενημερώνετε. Απλά ε, προσπαθώ να σε ενημερώσω εκ των προτέρων ε, ποιες τροπολογίες θα καταπέσουν εφόσον ψηφιστούν ορισμένες. Λοιπόν, προχωράμε στην ε, ψηφοφορία. Όπως ξέρετε, έχουμε την εισηγήτριά μας, την κυρία Γκυγιό, για το θέμα αυτής της έκθεσης, το οποίο είναι σε αναδιατύπωση, πρόκειται για τη διεθνή προστασία. Λοιπόν, τροπολογία υπαριθμών 5. Υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 80 είναι γλωσσικής φύσεως, 81 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Υπαριθμόν 6. Οι 82 και οι 83, μισό λεπτό, οι 60 και οι 82 είναι ταυτόσιμες. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 83. Όχι. 84. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 85, ε, μισό λεπτό, ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία υπαριθμών 7, λέει ο Πρόεδρος, και ε, ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 85 αποσύρθηκε, 86 υπέρ. Ε, εγκρίθηκε και αυτό, η 87 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Όχι, 88 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 89 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 92 και 93 ταυτόσιμες υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 94 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 9 υπέρ, να ελέγξουμε την 96. Εντάξει, ελέγχουμε την 96. Την 96 να ελέγχουμε, παρακαλώ, ε, ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. «29 υπέρ, 19 κατά, εγκρίνεται. Πάμε στην 9, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 97 προφορική τροπολογία της κυρίας ε, Φλότρ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε στην 10, τροπολογία 10. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ. Κατά αποχές. Νομίζω ότι απορρίφθηκε ε, να ελέγξουμε. 98 ελέγχουμε. Ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε για την 98, τώρα έκλεισε ψηφορία. 22 υπέρ, 26 κατά. Απορρίπτεται. Πάμε στην 99 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Ε, μισό λεπτό, 1.06 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 1.10 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 1.11 υπέρ κατά, ε, αποχές απορρίπτεται. Μισό λεπτό, νομίζω ότι απορρίφθηκε, λέει ο πρόεδρος. Ας ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 111, ε, 111. Ε, ελέγχουμε, ψηφίζουμε παρακαλώ. Εγκρίθηκε. Θέλετε να ελέγξουμε την 110. Ας ελέγξουμε την 110. Ε, Πάμε πίσω στην 110 παρακαλώ. 110. Ψηφίζουμε. Έκλεισε. Απορρίφθηκε. Πάμε στην 112. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 113 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 114 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Νομίζω ότι εγκρίθηκε. Κοιτάξτε, σα παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σα. Τα σηκώνετε κανονικά, τώρα μην αγκαζόμαστε να ελέγχουμε συνεχώ ηλεκτρονικά. Πάμε στην επόμενη. 114. Ε, Ψηφίζουμε. 114, παρακαλώ. Εντάξει, εγκρίθηκε. Η 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε και αυτή οι 15 και οι 118 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 και 119 και οι 120 ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά. Αποχέ συγκρίνεται. Και οι 121 υπέρ. Ε, για την 121 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 124 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 127 υπέρ. Για την 127 ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Νομίζω ότι εγκρίθηκε. Είδα ότι ψήφισαν μαζί η Φιλελεύθερη και το ΕΛΚ. Εγκρίθηκε. Να ελέγξουμε. Ας ελέγξουμε λοιπόν. Δεν θέλετε να ελέγξουμε. Λοιπόν, εντάξει. 129 υπέρ. 128 πρώτα. 128 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 129 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 130 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 131 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται όχι εγκρίθηκε έχετε δίκιο 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται οι 21 και 135 ταυτόσιμες υπέρ κατά εγκρίνεται. 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 140 υπέρ υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ, κατά, αποχέσει. εγκρίνεται. 141 υπέρ, κατά, Αποχέσει εγκρίνεται. Ελέγχουμε για την 141. Ψηφίζουμε λοιπόν για την 141. Έκλεισε η ψηφοφορία. Πράγματι απορρίφθηκε. Πάμε στην 142. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 143. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 144. Υπέρ. Κατά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 That's what I was saying. 152 does not fall. Ε, αυτό είπα ότι 152 δεν καταπίπτει. Αυτό είπα. Okay. Do we agree that 152 is falling too? Πιστεύετε ότι καταπίπτει και η 152. Εντάξει, τότε προχωράμε. Πάμε στην... Α, 178, στη σελίδα 10. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 179, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 180. Εγκρίθηκε 180, 26 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 181 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 182 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 183 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 184 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 έλεγχος για την 184 ελέγχουμε ή όχι για την 184 τι θα κάνουμε, θα ελέγξουμε, ελέγχουμε για την 184, ελέγχουμε, ελέγχουμε για την 184, ε, ψηφίζουμε, έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Τώρα, 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 185 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 186 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 187 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 188 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 και 189 είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 191 παρακαλώ. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 192 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 196 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 199 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 200 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 201 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μισό λεπτό, 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 202 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 203 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 204 υπέρ μισό λεπτό όχι όχι η 30 ψηφίζουμε για την 30. Όχι, πήγαμε στη 204. 204 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 205 και 206 από κοινού ε, υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 207 ελέγχουμε για την προηγούμενη 206 ελέγχουμε ηλεκτρονικά ε, και για την 205 είναι ψηφίσμα από κοινού. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. 2.07. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 208 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 209 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 210 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ο απορρίφθηκε Είχατε εντύπωση ότι υπερψηφίσατε. κανα λάθος. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. γιατί 210 ελέγχουμε. Ε, απορρίφθηκε. Το θέμα είναι να έχουμε συντονισμό χρονικό, πότε σηκώνεται το χέρι και πότε ψηφίζουμε για υπέρ ή κατά. Εν πάση λοιπόν, ε, για την 211 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 212 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Η 13 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 14 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 215 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Μάλιστα. 216 υπέρ υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 32 υπέρ Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Θέλετε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πολύ ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Εγκρίθηκε. 217 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 218 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 219 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές Νομίζω ότι απορρίφθηκε. 221 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. 222 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 225 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 34 αποσύρθηκε. 226 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 227 ελέγχουμε ε, ηλεκτρονικά την προηγούμενη παρακαλώ την 226 την ελέγχουμε ηλεκτρονικά ελέγχουμε έκλεισε η ψηφοφορία 28 έναντι 23 εγκρίνεται 227 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε στην 228 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 229 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 230 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 231 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 233 υπέρ. Νομίζω ότι η προηγούμενη εγκρίθηκε, λέει ο πρόεδρος. Νομίζω ότι εγκρίθηκε. 233 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 234 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 235 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 236 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 237 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 238 αποσύρεται. Η 36 υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται λάθος κάνει ο πρόεδρος το 239 ζητάει συγγνώμη 239 λοιπόν υπέρ 239 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 241 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ, κατά, αποχές ε, μισό λεπτό. Ψηφίζουμε πάλι Για την 38 παρακαλώ να σηκώσετε τα χέρια σας υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 40, 240 αποσύρθηκε, 242 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 39 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 243 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 244 καταπίπτει η 43 243 ελέγχουμε τη 243 έκλεισε η ψηφοφορία εγκρίνεται Τώρα περνάμε στην 244 καταπίπτει όμως αν δεν κάνω λάθος. Και περνάμε στην 249 και 250 ταυτόσημες. Ωραία. ψηφίζουμε από κενού. Υπέρ. Κατά. 249 και 250 από κοινού παρακαλώ. Να επαναλάβουμε. 249, 250 μαζί και οι δυο. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Η 43 καταπίπτει. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 253 υπέρ. 253 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. ε, 45. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 254 ε, υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται 255 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 256 απεσύρθη 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 και 257 ταυτόσημες υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 259. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 258. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 260. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 261. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 262 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 263 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 264 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά. εποχές. Εγκρίνεται. 265 υπέρ. Κατά. εποχές, Απορρίπτεται. 266 υπέρ. Κατά. εποχές, Απορρίπτεται. 49 υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται. Συμφαστική 10 υπέρ κατά παρακαλώ Πρόεδρε, όπως είπατε ήδη, ένα λεπτό, ένα λεπτό λοιπόν. Όπως είπατε ήδη, υπάρχει μια προφορική τροπολογία για τη συμβαστική 10 γιατί υπήρχε ένα σημαντικό πρόβλημα μετάφρασης του γερμανικού κειμένου. Συμφωνήσαμε με το τοξί του ΕΛΚ σοσιαλιστών ότι στον τίτλο θα διαγραφεί ο όρος ευρωπαϊκό και η πρώτη παράγραφος που δεν έχει πια κανένα νόημα και η τέος δεύτερη παράγραφος είναι τώρα η πρώτη παράγραφος και θα προσθεθεί στο F ε, ενέκρινε τις διατάξεις της συμφωνίας του Γενέβης χωρίς καμία γεωγραφική, κανένα γεωγραφικό περιορισμό. Αναφέρεται αναφορά δηλαδή συμφωνία της Γενέβης. Και μετά βέβαια η τεχνική προσαρμογή θα γίνει γιατί οι αριθμοί των παραγράφων μεταφέρονται. Αφού η πρώτη παράγραφος διαγράφεται. Αυτά. Πρώτα σας ευχαριστούμε κυρία Χίους για τις επεξηγήσεις αυτές, για την προφορική τροπολογία, για την συμβεστική τροπολογία 10. Το άρθρο 18. Ελπίζω όλοι να το σημειώσαν και μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία. Η κυρία Χολμαϊερ. Θα ήθελα να προσθέσω, Πρόεδρε, ότι η ψηφοφορία που κάναμε προηγουμένως για το άρθρο 33 ε, δεν θα χρειαζόταν να έχει γίνει λόγω του συμβασμού αυτού. Δεν θα χρειαζόταν δηλαδή να το έχουμε ψηφίσει αυτό. Γιατί αυτά που κάναμε αναφέρονταν στην ε, συμβαστική τροπολογία 10. Συμφωνείτε, συμφωνούμε όλοι. Κύριε Χίρς, συμφωνείτε. Ωραία. Περάμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Συμβιβαστική τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Αυτό σημαίνει ότι πολλές από τις τροπολογίες καταπίπτουν και περνάμε στην 271. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται νομίζω ναι ναι ναι απορρίφθηκε 272 απεσύρθη 273 κατά αποχές απορρίπτεται 274 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51 υπέρ Υπέρ, υπέρ, υπέρ. Υπέρ. Τις 51. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται, εγκρίνεται φαντάζομαι. Είδα αρκετά χέρια. Να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε. Έχουμε όλοι κουραστεί βέβαια. Αλλά αν δεν σηκώνουμε τα χέρια μας, δεν θα προχωρήσουμε. Χειρότερα είναι. Λοιπόν, να ελέγξουμε την 51. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 51. Πέρας. 28 προς 22. Ενεκρίθη λοιπόν πράγματι. 52 τώρα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 275 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 276 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 279 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 277 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 278 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 280 αποσύρθη 281 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 282. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 283. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 284. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 285. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 286 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Λογικές σκέψεις 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56 υπέρ κατά εγκρίνεται 57 υπέρ κατά εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 63. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 64. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 65. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66. Υπέρ. 66. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 67. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές δεν είδα κανένα χέρι να σηκώνεται. Λοιπόν, 76. Παρακαλώ. 76. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 77. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4 και 78. Ταυτόσημες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι είναι κρίμα. Και 79. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία του κειμένου. Α, όχι ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Φαίνεται ότι ξέχασα δύο. Καθοδόν τις έχασα. Είστε σίγουροι. Είστε σίγουροι δύο. Λοιπόν. Σελίδα 17. Δύο τροπολογίε. Σελίδα 17 ψηφίζουμε 251 και 252 ταυτόσημες. Και οι δύο ταυτόσημες σελίδα 17. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. Και τροπολογία 44. 44. Πάντα σελίδα 17. Η 44 υπέρ. Ναι, 44 βλέπω εγώ εδώ. 43 ψηφίσαμε ίσως. Όχι. Ανάποδα. Δεν ψηφίσαμε 43. 43 λοιπόν. Καταπίπτει. Ωραία. Η 44 τότε. I've been told that it was not voted. Μα μου είπαν ότι δεν ψηφίστηκε. Ακόμα και η τεχνική υπηρεσία μπορεί να κάνει ένα σφάλμα, αλλά μου είπαν ότι λείπει αυτή η ψηφοφορία. Όχι, ψηφίσαμε. Ωραία, εντάξει. Τελειώσαμε λοιπόν. Και περνάμε στην τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά για το σύνολο του κειμένου ω τροποποιήθηκε. Ψηφίζουμε τώρα, έχει την ψηφοφορία. Now the vote is closed. Πέρασε τη ψηφοφορία. 28 υπέρ, 22 κατά. Συγχαρητήρια κύριε Γιλιόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ε, κυρία Λάτφορντ, ένα, ένα λεπτό. Εγώ είμαι κάποιος που δεν έχει πολύ υπομονή. Μήπως οι συντονιστές μπορεί να εξτάσουν το θέμα της ψηφοφορίας. Περάσαμε πάνω από δύο ώρες με την ψηφοφορία αυτή. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο. Δεν ήταν ίσως τόσο εύκολο όσο σε άλλες ε, ψηφορές να προχωρήσουν με τις, ε, ε, με τις συμβαστικές τροπολογίες. Δεν μπορεί να γίνει όσο δουλειά που έγινε από την κυρία Σίπελ για συμβαστικές τροπολογίες, αλλά εάν υπάρχει δυνατότητα, δεν ξέρω. Δεν επιτρέπεται δύο ώρες και ένα τέταρτο να ψηφίζουμε. Πρόεδρο, το μόνο που μπορώ να συμφωνήσω μαζί σα είναι ότι η υπομονή ποτέ, ποτέ δεν ήταν οι μα μου Δεύτερον, κάνω ό,τι μπορώ για να επιταχύνω. Αλλά σας λέω, καμιά φορά έχουμε πολύ χρονοβόρες διαδικασίες. Όλοι θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε. Τι να γίνει. Η Επιτροπή ΛΥΜΕ έτσι φαίνεται ότι λειτουργεί. Περνάμε από αυτές τις ε, μαζικές πληροφορίες, όχι που και που, αλλά συχνά. Όλες οι άλλες επιτροπές ε, του σώματος εδώ δεν το έχουν αυτό. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την απόδοση των συντονιστών και των μελών της ε, Επιτροπής μας στην Πληροφορία. Κύριος Μωράης. Κοιτάξτε. Ε... Ήταν πολύ καλή η ψηφοφορία αυτή σήμερα. Σας συγχαίρω. Σας ευχαριστώ και στην εργασία σας, κύριε ο Πρόεδρος again at 3 p.m. this afternoon. Τρεις το απόγευμα ξαναβρισκόμαστε.